την ημερήσια διάταξη. Το τελικό σχέδιο της ημερήσια διάταξη όπως εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των πρέδρων στις 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 149 του κανονισμού, έχει διανεμηθεί. Δεν έχω λάβει καμία πρόταση τροποποίησης ημερήσια διάταξη. Επομένω, αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, κάποιο αίτημα τροποποίηση, η ημερήσια διάταξη θεωρείται επομένω εγκριθήσα.